Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίσω την έναρξη της σημερινής συνόδου. Καλή μας ημέρα. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, έκθεση Χάουταλα επί της ετήσιας έκθεσης